του φασισμού του γνήσιου παιδιού της καπιταλιστικής βαρβαρότητας αυτής που όλοι σας υπερασπίζεστε. Η ιστορική αλήθεια, η κόκκινη σημαία στο Reichstag αποτελούν άσβεστο μάρτυρα το ποιο εξολόθρεψε τον ναζισμό, το ποιο θρέφει και σήμερα την ακροδεξιά, τον εθνικισμό, τους φασίστες, το μαρτυρά το τι γίνεται σήμερα στην Πολωνία, την Ουγγαρία, τις Βαλτικές χώρες με τις διώξεις και απαγορεύσεις κομμουνιστικών κομμάτων την ίδια ώρα που απονέμονται τιμές σε συνεργάτες των Ναζί με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσα ιδρύματα ψέματα στα σχολικά βιβλία και ακριβοπληρωμένε καμπάνιες και αν χρηματοδοτήσετε την ιστορία τη γράψανε και τη γράφουν οι λαοί με την πάλη του ενάντια στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Είναι ιστορικές κατακτήσεις του σοσιαλισμού σε παιδεία, υγεία, εξάλληψη της ανεργίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καπιταλισμός δεν είναι μονόδρομος. Οι λαοί μπορούν με τη δική τους εξουσία στις χώρε του να παλέψουν για την Ευρώπη του σοσιαλισμού. λεπτό ο ε, ολοκληρωτισμός είναι κατά των ελεύθερων δικαιωμάτων, ε, καταπίεση, ε, βιότητες. Αυτό αυτά ήταν αυτά που συνέβαιναν στα απολυταρχικά καθεστώτα. Για πάρα πολλά χρόνια αυτή ήταν η ιστορία στην Ευρώπη. Και ευτυχώ, ε, ελπίζω και για το μέλλον, να μην ξαναυπάρξουν τέτοιου είδου καταστάσει. Για να μην υπάρξει όμω κάτι τέτοιο που δεν είναι στο μέλλον, δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό το κομμάτι τη ιστορία. Πρέπει να διατηρούμε ζωντανή τη μνήμη στον φασισμό, τον ναζισμό, αλλά και στα απολυταρχικά κομμουνιστικά καθεστώτα. Και αυτό πρέπει να παραμείνει στη συνείδηση των λαών. Γι' αυτό λοιπόν να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα πολιταρχικά καθεστώτα, τις επιπτώσεις τους στη ζωή των ανθρώπων, ε, τις επιπτώσεις στην παιδεία, να έχουμε μια σωστή παιδεία για να μην ξεχάσουμε ε, πολλά πράγματα. Σημαντικά είναι και τα πανεπιστήμια. Εμείς φέρουμε την ευθύνη για τις μελλοντικέ γενναίες, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν καταστάσεις, έτσι ώστε να μην επανεμφανιστεί ο ε, απολυταρχισμός στην Ευρώπη. Η κυρία Κώστα παρακαλώ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι το δημοκρατικό πρόγραμμα της αλληλεγγύης ε, δεν μπορεί να βασίζεται στην άγνοια της κοινή μας ιστορικής, ε, της κοινής, ε, του κοινού παρελθόντος. Ποτέ πια να μην υπάρχει απολυταρχισμός, ποτέ πια ολοκαυτώματα να σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιεπρέπεια. Μπροστά λοιπόν στους νέους κινδύνους των εθνικισμών, των ρατσισμών, αλλά και μπροστά στον ρεβιζιονισμό και στον αρνητισμό, είναι απαραίτητο να έχουμε μια νέα παιδεία στην Ευρώπη η οποία θα λαμβάνει υπόψη της ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει έρευνα στην ιστορία, κοινή μέθοδος, ε, κοινή διδασκαλία της ιστορίας μέσα από κοινέ σπουδέ ε, κριτικές προσεγγίσεις για να υπάρξει πραγματική επανένωση της Ευρώπης. Πρέπει βεβαίως και να εξοικειωθούμε και με τη μυθολογία γιατί θεωρώ ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να φτάσουμε και στο ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας πυρήνας κοινό στην ιστορία της Ευρώπης ε, το οποίο θα βρίσκεται και στη βάση της ε, ενοποίησης. Δεν αρκεί βέβαια να έχουμε μόνο τη μνήμη για να μπορούμε να αποφύγουμε κινδύνους γνωρίζουμε ότι ακόμα και αν υπάρχουν όλα αυτά ε, θα πρέπει να έχουμε πιο κριτική άποψη και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο αν δεν υπάρχει συνείδηση. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι δεν φτάνει να καλλιεργούμε μόνο τη μνήμη, αλλά να έχουμε και μια δημοκρατική συνείδηση η οποία ε, ξεπηδάει από αυτό το ποτέ πια το ποιου που οδήγησε στο να υπάρχει το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Υπήρξαν ε, ενδιαφέροντα θέματα αλλά και αρνητικέ εξελίξει στα σχολεία. Υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε που προσπάθησαν στα ιστορικά σχολεία να ε, συμπεριλάβουν την ιστορία του ολοκαυτώματο, ε, σήμερα στην Τσεχία όμως ε, μερικοί αντί να ε, αναφέρονται στο Γιάν Πάλακ ούτε και στην Ουγγαρία πολλοί αναφέρονται που θα έπρεπε να αναφερθούν. Ρεβιζιονισμός λοιπόν ως προς τους ήρωες. Γι' αυτό ας προσπαθήσουμε να βασιστούμε στις θετικές μας εμπειρίες. Uh, uh, Κυρία Σολέ, ένα λεπτό Κύριο Σολέ, συγγνώμη. Είμαστε στην εποχή της μεταλήθειας, των fake news. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Θα πρέπει να θωρακιστούμε με παιδεία, με μέσα επικοινωνίας πλουραλιστικά. Θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι, πεπαιδευμένοι οι πολίτες. Και έτσι θα αντιμετωπίσουν αυτούς που θέλουν να χαλκεύσουν την ε, ιστορία. Όπως ο Παύλο Κασάδο του Λαϊκού κόμματο που λέει ότι οι Ισπανοί δεν έκαναν ε, απικίες αλλά προσπάθησαν απλώς να μεγαλώσουν την Ισπανία αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την προσβολή στην μνήμη, να την διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη για αυτούς που δεν μπόρεσαν να έχουν δημόσιο βήμα, να μην έχουμε ένα κομμάτι ιστορίας που είναι ξεχασμένο δικαιοσύνη και αποκατάσταση αυτών που αδικήθηκαν. Και αυτά όχι μόνο με την μνήμη των φρικαλαιοτήτων, των ολοκληρωτικών καθεστώτων, αλλά όλων των καθεστώτων που βάσισαν την εξουσία ε, πατώντας επί της παραβίας των δικαιωμάτων. Ρουμπάν Κρέσπο είναι ο επόμενος, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η Ισπανία είναι μια εξαίρεση στην ε, Ευρώπη, γιατί υπάρχει ατιμορρησία. Έχουμε μνημεία που παραπέμπουν στη δικτατορία του Φράγκο. Μόνο στην Ισπανία έχουμε κάποια νομικά πρόσωπα που επιδοτούνται και παραπέμπουν ε, σε γενοκτονίες, σε φασισμό, γιατί έχουμε χιλιάδες ε, πτώματα τα οποία είναι ε, σε, σε ομαδικούς τάφους και τους έχουμε βγάλει. Μόνο στην Καμπότζη έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Κοιτάξτε τι έγινε στην Αργεντινή και εκεί έγιναν κάποιες ε, έρευνες τόσο ώστε να πάνε στην δικαιοσύνη κάποιοι που εγκλημάτισαν κατά της ανθρωπότητας και ήρθε ο Επίτροπος Τίμερμανς και είπε για τα θύματα, είπε για τις οικογένειές τους αλλά δεν έγινε τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να συνεχίσει να, αδρανά, να δρανεί ενώπιον των θυμάτων του φραγκισμού αλλιώς είναι συνένοχος σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος Πρέτσελ ένα λεπτό Αξιότιμε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν πρόκειται για την μνήμη στα ε, σοσιαλιστικά και εθνικοσοσιαλιστικά καθεστώτα του προηγούμενου αιώνα, ε, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει τα ιστορικά βιβλία να διδάσκουν για όλα αυτά. Όταν όμω πρόκειται για το να ζητήσουμε κοινέ αξίε, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Γιατί στο θέμα τη σχέση ανάμεσα στο εθνικό κράτο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί υπάρχουν συζητήσει για αυτέ τι αξίε και είναι πολύ καλό που γίνονται αυτέ στις συζητήσεις και με ανοιχτό ε, κάθε ενδεχόμενο. Το θέμα δεν είναι να αποδίδει κανεί σημασία μόνο στο, στην κοινότητα, αλλά και στο άτομο. Δεν πρόκειται μόνο για την ευρωπαϊκή διάσταση. Ούτε καν πρόκειται για τη μία και μόνη αλήθεια. Πρόκειται για ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα οποία αυτά μόνο μιλάνε για τη μία και μόνη αλήθεια. Για να αποκτήσει κανεί την αλήθεια πρέπει να αγωνιστεί, να υπάρχει παιδεία, αλλά δεν είναι δουλειά των κρατικών θεσμών να εκπαιδεύουν αυτό το κάνουν μόνο τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Και νομίζω κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να απέχει, μακρά να απέχει από όλα αυτά τέτοιου είδου προσπάθειε. Ο κύριο Λαμασούρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαίρω τον συνάδελφο Κοβατσέκ που είχε την πρωτοβουλία για τη συζήτηση αυτή. Δεν είναι ε, κοινωτική αρμοδιότητα η εκπαίδευση και δεν πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να φροντίσει να μην επανεμφανιστεί πουθενά στην Ευρώπη ε, ένα λόγο που θα είναι λόγο μίσου στην Ευρώπη. Σε δύο γενιέ πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ε, καταστροφή του πολέμου στη σχεδόν διαρκή ειρήνη. Και αυτό ήταν ένα θαύμα το οποίο κατέστη δυνατό μόνο χάρη στη δημιουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που χρόνο με το χρόνο συμφιλίωσε του λαού χωρί να του στρέφει τον έναν εναντίον του άλλου, αλλά όλου του ε, συνένωσε γύρω από ένα κοινό σχέδιο ολοκλήρωση της Ευρώπη. Με τα παιδιά μα, λοιπόν τώρα καταλήγουμε να φτιάχνουμε μια καινούργια γενιά εθνικιστών, μιλώντας για fake news, ε, αρνούμενοι της, ε, την ιστορία και τις τραγωδίες του 20ου πολέμου, δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε κάποια εθνικά αφηγήματα, αλλά πρέπει να έχουμε εθνική ιστορία. Κυρία Λιμπάτσκα, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Τα πολιταρχικά καθεστώτα είναι ένας πολιτισμός βίας. Αρνούνται την ελευθερία της σκέψης. Η μνήμη, λοιπόν, είναι σημαντική. Η μνήμη των εθνών και της ηρωικής συμπεριφοράς των πολιτών. Τα τωρινά πολιταρχικά συστήματα συχνά παρουσιάζονται ως δημοκρατικά καθεστώτα και αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο γιατί μας κάνουν να εφησυχάζουμε και γι' αυτό καθήκον μας είναι να εκπαιδεύουμε τους νέους ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον κόσμο με κριτική σκέψη, να κατανοούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να συνεργάζονται με άλλους με ανεκτικότητα και σεβασμό προς τους άλλους. Η εκπαίδευση είναι το πιο αποτελεσματικό στοιχείο για την καταπολέμηση του μίσους, της μυσαλλοδοξίας και του απολυταρχισμού. Τα λόγια της Ίντιρα ε, Γκάντι απεδείχθησαν αληθή ήταν, έπεσε θύμα μίσους και εκείνη. Δεν θέλουμε να είμαστε ε, μαθητές του μίσους. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριο Τάραντ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Τζον Ντάν είπε μη ρωτά για ποιον χτυπάει η καμπάνα, η καμπάνα χτυπάει για σένα, όπως είπε και παραφράζοντας τον Hemingway απολυταρχισμός μπορεί να έχει πολλά χρώματα, να είναι αριστεράς, δεξιάς, νατσιστικός, τροτσχιστικός, οτιδήποτε. Σημαντικό είναι ότι πρέπει να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον απολυταρχισμό και να τον αντιμετωπίσουμε όταν είναι ακόμη στο στάδιο του σπόρου και πριν να γίνει ε, ένα τεράστιο δένδρο. Πριν από ένα μήνα δημοσιεύθηκε ένα βιβλίο από ένα εσθονό συγγραφέα που ξέρει πώς να αναγνωρίζει τον απολυταρχισμό. Λέγεται Ένζαρ, ήταν φυλακισμένος ε, στο Στούτσχοφ, γιατί ήταν εχθρός ε, του Γερμανικού Ράι και αργότερα ήταν και στο Γκουλάγ, γιατί ήταν και εχθρός των Σοβιετικών. Διδάχθηκα πολλά από αυτόν και ελπίζω με αυτό το ένα λεπτό παρέμβασης να σας δίδαξα κι εγώ κάτι. Κυρία Φορέντζα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω τώρα εδώ χρόνο για να τοποθετηθώ στο ρεβιζιονισμό που φάνηκε σε αρκετές ε, παρεμβάσεις. Στις 9 Μαρτίου γίνονται γιορτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχνάμε ότι υπάρχει και η νίκη του ερθρού ε, στρατού κατά του ναζισμού Θέλω λοιπόν να πω ότι εγώ είμαι πολύ περήφανη που μπόρεσα και εγώ εδώ να συμβάλλω στο ότι υπήρξε ένα ψήφισμα ε, όπου απαγορεύονται όλα τα νεοφασιστικές οργανώσεις. Ε, ε, θα πρέπει να συλλαμβάνονται αυτοί οι φασίστες. Συνέβη αυτό στο Μπάρι και εδώ πρέπει να μην ξεχνάμε ποια, ποιες είναι οι ρίζες του πολιταρχισμού και στην Ιταλία και στην Ευρώπη. 49 άτομα μένουν στη θάλασσα χωρίς να θεωρούν καν άτομα. Όταν δημοσιεύεται η σύλληψη ενός ανθρώπου όπως του Τσέζαρε Μπατίστη βρισκόμαστε σε απάνθρωπες εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη μιλήτρια, ε, κυρία Σόιντροβα, για ένα λεπτό. <coughs> Συνάδελφοι, το να ε, διδάσκει κανείς τον ε, ολοκληρωτισμό, αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν ε, θέλω να σας παραπέμψω σε ένα τσέχικο πρόγραμμα, το Post Bellum. Είναι μια οργάνωση η οποία συγκεντρώνει αναμνήσεις από ανθρώπους που θυμούνται εκείνη την εποχή και αυτά τα περνάνε μετά στα σχολεία. Ε, το κλειδί είναι οι δάσκαλοι. Πρέπει να τους στηρίζουμε και να τους δίνουμε όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούμε. Γι' αυτό έχουμε ε, το βραβείο Γιάνν Άνος για τους δασκάλους. Αυτό το στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να ξεκινήσει εφέτος. Αυτή θα είναι η δική μας συνεισφορά προς εκείνους τους εκπαιδευτές που ενημερώνουν τους πολίτες και το σπίτι της ευρωπαϊκής ιστορίας που το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στις 20 Μαρτίου ε, θα υπάρξει μια έρευνα για τον Γιάν Παλάχ ε, τον οποίο τον έχουν ήδη προναφέρει αρκετοί. Πολύ ωραία. Επόμενη ομιλήτρια, ε, Ροντρίγκε, ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όπως είπαμε, αυτή η συζήτηση ε, που λαμβάνει η χώρα θα πρέπει να ασχοληθεί με τα, με τα χειρότερα δικτατορικά καθεστώτα και αριστερά και δεξιά. Ε, τώρα δεν πρόκειται για, την, για τον ιδεολογικό προσανατολισμό. Υπήρξαν δικτατορίες ε, στην Ευρώπη, αλλά οι δικτατορίες αυτές συγκαλύπτονται, εμφανίζονται ως δημοκρατίες και ελεύθερες κοινωνίες. Ε, χρησιμοποιούν μια γλώσσα για να παραπλανήσουν τους ε, πολίτες. Και νομίζω αυτό θα πρέπει να αρκεί για να ντρέπεται κανείς, διότι πάρα πολλοί ε, πέθαναν για να αντιμετωπίσουν τον ολοκληρωτισμό και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο χρειαζόμαστε την παιδεία. Να μην ξεχνάμε τον Έλιοτ, αυτά που είπε ο Έλιοτ όπου ανέφερε ότι θα πρέπει κανείς όλοι να μάθουν από την ιστορία και δεν θα ξέρουν γιατί ακριβώς πράγμα μιλάω. Ο κύριος Κέλαμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πριν από 10 χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν θα είναι πραγματικά ενωμένη εάν δεν μπορέσει να επανενώσει την ιστορία της, να συμφιλιώσει τις έννοιες ε, αναγνωρίζοντας ότι ο κομμουνισμός και ο ναζισμός ε, έχουν ένα, είναι ένα παρελθόν εγκλημάτων. Ε, εορτάζουμε την επέτειο από την ανέγερση, από την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Παρ' αυτά, Χρειάζεται ε, μια διεθνής δέσμευση, η οποία θα είναι συνεχής και χρειάζεται να υπάρχει επίγνωση των πολιτών για όσα συνέβησαν στην Ανατολική Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι γνώσει για το θέμα αυτό δεν είναι ακόμη επαρκή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε για το τι πρέπει να γίνει και υπενθυμίζω κάποια από τα σημεία που είχαν αναφερθεί. Δημόσια συζήτηση για το, τα απολυταρχικά συστήματα, ε, επικαιροποίηση των σχολικών βιβλίων ιστορίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να συντονίσει αυτό το έργο, πιστεύω. Και η 23η Αυγούστου να οριστεί η μέρα μνήμης για όλα τα θύματα του απολυταρχισμού. Ευχαριστώ. Κυρία Ward, ένα λεπτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε ως ε, ένα σχέδιο ειρηνευτικό μετά τις ε, φρικαλαιότητες του παρελθόντος. Πέρυσι, το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς προώθησε τον κοινωνικό διάλογο και έδωσε τη δυνατότητα σε 6 εκατομμύρια ε, άτομα να λάβουν ε, μέρος σε εκδηλώσεις στις, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ενισχύσουμε την πολυμορφία μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευση για όλες τις ηλικίε θα πρέπει να διδάσκουμε την ιστορία καθώς και τα εξαιρετικά επιτεύγματα. Υπάρχουν πολλές δύσκολες στιγμές του παρελθόντος μας που πρέπει να τις αναγνωρίσουμε και πρέπει να τις διδάσκουμε στα σχολεία μας. Η γενοκτονία των Ρωμά, η ένδια στην Ολυμό στην Ουκρανία που οδήγησε στο θάνατο ε, 7,2 εκατομμυρίων ατόμων. Θα πρέπει οι λαοί τη Ευρώπης να διδαχθούν από τα σφάλματα του παρελθόντος και να συνεργαστούν. Όπως είπε η κυρία Μέρκελ, πρέπει οι γενιές να επιβιώσουν μετά τον πόλεμο. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σας διακόπτω για να τηρούμε το χρόνο. Γουόγκα, ένα λεπτό. Και προσωπικά είχα να αντιμετωπίσω το, το ότι ε, δεν υπάρχει μνήμη του απολυταρχικού καθεστώτος ε, του παρελθόντος. Κάποιο έγραψε μια επιστολή στο Jeff Bezos, ε, του CEO του Amazon, να αφαιρέσει κάποια σοβιετικά σύμβολα. Και μου έκανε εντύπωση, μου έκανε κάποιες αντιδράσεις άλλων ευρωβουλευτών που δεν είχαν συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό ήταν αυτό και πόσο σημαντικές ε, ήταν οι φρακαλαιότητες του σοβιετικού καθεστώτος. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για σουβενίρ όταν μιλάμε για το σφυροδρέπανο Σκοτώθηκαν εκατομμύρια, εξορίστηκαν εκατομμύρια. Η βία του σοβιετικού καθεστώτος υπολογίζεται ότι είχε περίπου 60 εκατομμύρια θύματα. Ο υπόλοιπος κόσμος λίγα ήξερε για το τι γίνεται πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα θα πρέπει τα κομμουνιστικά σύμβολα να τα αντιμετωπίσουμε λίγο πολύ όπως αντιμετωπίζουμε και τα ναζιστικά σύμβολα. κύριος Νέκοφ, ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, η ιστορική μνήμη για το ολοκληρωτικό παρελθόν είναι κάτι που θα πρέπει με προσοχή να το προσεγγίσουμε και έτσι λόγω του χρόνου με μεγαλύτερη ψυχραιμία, αποστασιοποιημένη, γιατί είδαμε τι έγινε στο πρώην κομμουνιστικό μπλοκ. Εκεί, ξέρετε, ακόμα μνήμες είναι ζωντανές. Ε, Πρέπει στο σχολείο να ενημερωθεί καινούργια γενιά. Χρειάζεται μια τέτοια ιστορική προσέγγιση να είναι αντικειμενική. Στα πρόσφατα σχολικά βιβλία ο κομμουνισμός περιγράφεται ως το χείριστο δυνατό φαινόμενο. Όμως, πολλοί νοσταλγούν τις εποχές εκείνες, διότι κατά την ε, μετάβαση στη δημοκρατία οι άνθρωποι στριμώχτηκαν, δυσκολεύτηκαν. Δεν θα πρέπει να έχουμε μανιχαϊσμό, κομμουνισμό, αντιμηχανισμό. Θα πρέπει να ποντάρουμε στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Την ένταξη. Ευχαριστώ. Και τώρα, η Επίτροπος σας λαβεί το λόγο για να απαντήσει. Λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ενδώσω στον περισμό να την ε, μητρική μου γλώσσα. Γιατί έχουμε σήμερα την πεντηκοστή επέτειο ενός φοιτητή που αυτοπυρπολήθηκε στο Πανεπιστήμιο της Πράγας με τη σημερινή συζήτηση συνειδητοποιούμε πόσο συμβολικότητα υψηλή έχουν αυτά σε σχέση με την μνήμη του ολοκληρωτικού παρελθόντος σε σχέση με τις λογοκρισίες. Ήμουνα σχεδόν 15 και η μητέρα μου μου είπε στο αυτή ποιος ήταν ο Πάλαχ που αυτοπεριπολήθηκε και τι έγινε ακριβώς το 69. Τα θυμάμαι πάρα πολύ ζωντανά αυτά. Και τι μου είπε, μην ξαναπείς ποτέ αυτό το όνομα, αλλά και να μην το ξεχάσεις. Πάμε στον Ιανουάριο του 89. Και τότε, τότε στην ε, πρατεία Βέντσεσλας, στην Πράγα, αυτό ήταν το σύνθημα. Το όνομά του που ήταν σύνθημά μας. Δεν πήγε χαμένη η θυσία του εξυπηρέτησε έναν ιστορικό σκοπό στην Τσεχοσλοβακία. Και σήμερα είναι ζωντανή η μνήμη του και στην Τσεχία και παντού. Γιατί θυμόμαστε ότι αυτά τα κατεστώτα φέρνουν καταστολή, λογοκρισία, φέρνουν μετανάστευση, φέρνουν καταράκωση της ηθικής και των ηθών. Γι' αυτό δεν πρέπει να ξαναγυρίσουν. Τώρα όσον αφορά την παιδεία, δεν νομίζω ότι κανεί σήμερα ή κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα να δίνει μία και μοναδική αλήθεια, μαθαίνει μοναδική αλήθεια στα παιδιά. Γιατί αυτό είναι ο ολοκληρωτισμό. Θέλουμε να υπάρχει αμεροληψία στην ιστορία στα σχολεία. Να διδάσκουμε τη νέα γενιά, να ξέρουν τι πληροφορίε, να έχουν κριτικό πνεύμα, διότι αν κανείς πιστεύει ότι μόνο τα σχολεία θα εξασφαλίσουν την γνώση της ιστορίας, αυτό θα ήταν πάρα πολύ αφελές. Σήμερα υπάρχει το ίντερνετ. Όπως είπατε, υπάρχει εκτεταμένη παραπληροφόρηση. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να ενημερώσουμε τους νέους, να τους μάθουμε πώς να ψάχνουν τις πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται μετά. Νομίζω ότι αυτό είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθήκον των κρατών μελών. Συνήθως εμπιστεύομαι τα κρατημέλη. Θεωρώ ότι δεν θα επιτρέψουν να κατησχίσει ολοκληρωτισμό στην παιδεία μας. Ο πρόεδρος λυπάμαι, λέει ο πρόεδρος γιατί ανησυχούν πολλοί συνάδελφοι που δεν θέλουν προπαγάνδα αλλά δεν κάθισαν να ακούσουν την γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, εκ μέρους του Συμβουλίου. Κύριε Σιώτη, σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική, δημιουργική αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση. Πόσο σημαντική είναι η παιδεία για να φτιάξουμε μια Ευρώπη κοινών αξιών αμοιβαία κατανόησης των παραδοσιών μας της ευρωπαϊκής ιστορίας και συμπεριλαμβανομένου του ολοκληρωτισμού. Να είστε σίγουροι στο κοινοβολίο ότι εμείς αυτό το θέμα θα το θεωρούμε υψηλή προτεραιότητας και στο μέλλον. Και πάλι σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος, πέρα τη συζητήσεως. Το επόμενο θέμα μας είναι έκθεση Τέρι Κάμπρας. Κατάσταση θεμελιδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017. Έχει τον λόγο εισηγητής για τέσσερα λεπτά. is yours, Rapporteur. Oh, you. Thank you. President, Commissioner and colleagues. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι και εσείς οι σκιώδεις εισηγητές για αυτήν την ετήσια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017 η έκθεση θα έπρεπε να είναι σχετικά σύντομη και το καταφέραμε. Θα έπρεπε κανεί να λάβει υπόψη όλα τα δικαιώματα ε, για το 17 στην Ένωση. Είναι σαφέ ότι κανεί μπαίνει σε πειρασμό να πει πάρα πράγματα. Αυτό το αποφύγαμε. Επικεντρωθήκαμε σε έξι βασικά θέματα. Μερικά από αυτά βέβαια ε, απασχολούν περισσότερο όγκο σελίδων ε, γιατί μας απασχολούν. Ε, μετανάστευση, γυναίκες, ε, κράτος δικαίου, ΜΜΕ, ελευθερία έκφρασης, ε, όχι στην ξενοφοβία, όχι στην ρητορική του μίσους και έτσι είπαμε ότι και συμφωνήσαμε την πρώτη στιγμή όσον αφορά τα κριτήρια πώς θα πρέπει να δουλέψουμε και τα βασικά μας κριτήρια είναι η κοινή μας πεποίθηση ότι δεν θέλουμε να έχουμε μια τελείως ουδέτερη ανάλυση. Ο στόχος μας ήταν να έχουμε μια, ένα κοινό προβληματισμό για αυτές τις βασικές αξίες. Όχι μόνο τις ε, προασπίσουμε, αλλά και να προτείνουμε πώς μπορούμε να έχουμε τη βελτίωση του χάρτη των δικαιωμάτων. Προσωπική παρατήρηση. Κανείς δεν πιστεύει ότι ο χάρτης θα είναι καλύτερος εάν παραμείνει το άρθρου 51. Αυτό θα πρέπει να ερμηνευτεί έτσι, ούτω ώστε να πρέπει να προχωρήσουμε και να σπεύσουμε βραδέως. Γι' αυτό σας λέω, έχουμε αναδείξει κάποια συγκεκριμένα ζητήματα για το κράτος δικαίου. Τονίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικότητα για τις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2. Αλλιώς αυτό υπονομεύει την εμπιστοσύνη, την αξιοπιστία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μετανάστευση μας προβληματίζει ακόμα. Το 2017 είχαμε 650.000 που ζήτησαν διεθνή προστασία και άσυλο στα κατημέλη για πρώτη φορά. Και πάνω από Χίλιοι πρόσφυγες πνίγηκαν στην Μεσόγειο. Ανθρωπιστική βοήθεια ποινικοποιήθηκε. Τα κράτη δεν μπόρεσαν να λύσουν τον κόριο δεσμό της κατάλληλης νομοθεσίας. Όλα αυτά τα λέμε στο κείμενο, γιατί τώρα για κάποιες χώρες, κάποιοι άνθρωποι ε, δεν τα έχουν χωνέψει αυτά. Ελευθερία της έκφρασης, μη ελευθερία του συνέρχεστε, ήταν πάντα ένα πρόβλημα αλλά και η ελευθερία τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να θωρακιστούν ακόμα και σε χώρες που δεν το περιμένει κανείς απειλούνται αυτά τα δικαιώματα. και πολλοί ακτιβιστές ε, κινδυνεύουν, ρατσισμός, ξενοφοβία, ρητορική μίσους, ε, έλλειψη ανεκτικότητας, όλα αυτά θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία των ανθρώπων. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που να αρνούνται την ανεκτικότητα, να φέρνουν διάκριση, δυσμενή. Μα θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, θα πρέπει να υπάρχει έτσι κατάλληλη ατμόσφαιρα. Εν κατακλείδη, μιλήσαμε για την ΦΡΑ, την, τον φορέα για τα δικαιώματα. Ε, το έργο που επιτελεί είναι εξαιρετικό. Ποτέ άλλο δεν το είχαμε πει η ΦΡΑ θα πρέπει να αναπτύξει δραστηριότητα όχι μόνο όταν τη ζητείτε, θα πρέπει να ενεργεί με ίδια πρωτοβουλία σε κάθε περίπτωση που διακυβεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ή καταπατούνται. Νέα εντολή χρειάζεται. Αυτές οι 21 σελίδες αποτελούν ένα κείμενο, κατά τη γνώμη μου, ένα κείμενο που είναι σαφές ε, και παραγωγικό. Ευχαριστούμε όλους και τους συμβούλους μας όλοι βοήθησαν ούτως ώστε να έχουμε αυτό το ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας ε, κυρίες και κύριοι. Και τώρα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να τηρείτε το χρόνο ε, που προβλέπετε για σας, ε, γιατί στις 5 ώρα θα αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Αν μιλάτε, μιλήσετε πάρα πολύ θα πρέπει να σας ε, διακόψω. Τώρα, ε, κύριε Επίτροπε, σας δίνω το λόγο. κύριε Γιούροβα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ότι εστιάζεται στα ε, θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξεκινώ με την νομοθεσία που είναι πολύ σημαντική για την ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια δεσμεύεται στο να επιβάλλει το κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική και ελέγχεται και η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Ε, το κράτος δικαίου ποτέ δεν ήταν τόσο καλά θωρακισμένο και ποτέ δεν ήταν τόσο ψηλά στις προτεραιότητές μας όπως σήμερα. Η Επιτροπή προτείνει μια τροποποίηση για την προστασία του ε, προεπιλογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν εντοπιστούν κάποια, κάποιες ελλείψεις στο κράτος δικαίου στα κράτη-μέλη. Και η Κομισιόν θέλει να αναλάβει πρωτοβουλίες για να ενισχύσει περαιτέρω το κράτος δικαίου, ε, υπόψη τη δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του ψηφίσματος <clears throat> για το μηχανισμό του κράτους δικαίου που εγκρίθηκε το 2016, όπως επίσης και τις συζητήσεις που ακολούθησαν. Μετά από τις ενέργειες της κυβέρνησης της Πολωνίας, ε, δρομολογήσαμε τη διαδικασία άρθρο 7 και το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους το Κοινοβούλιο αποφάσισε να δρομολογήσει την ίδια διαδικασία μετά από τις ενέργειες της Ουγγρικής κυβέρνησης. Πρόκειται λοιπόν για ε, πρωτοφανή βήματα και επίση η Επιτροπή χρησιμοποιεί και τη διαδικασία επιπαραβάση για να αντιμετωπιστούν διάφορες παραβάσει Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από πλευρά κρατών μελών. Χρησιμοποιούμε και άλλα εργαλεία, ελέγχου, έρευνε που έχουν σχέση με τη χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και άλλα εργαλεία που προβλέπονται στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σε γενικές γραμμές, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα του δικού της του συστήματος δικαιοσύνης. Οι εθνικοί δικαστές είναι και δικαστές της Ένωσης. Ε, βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό, μαζί μάλλον με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είναι οι θεματοφύλακες της τάξης, της ευρωπαϊκής, κυρίως ε, του ρόλου ε, που ε, μπορεί να παίξουν αυτοί οι θεσμοί στην προδικαστική διαδικασία. Να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις δικαστικές αρχές και αυτό αναφέρεται στην τελευταία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπου επισημαίνεται ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι καθοριστική σημασία για να υπάρχει ουσιαστική δικαστική προστασία. Σε τελική ανάλυση ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε πρόσφατα ότι η αποτελεσματικότητα αποτελεσματική προστασία είναι μία από τις αξίες ε, πάνω στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, θέλω να υπογραμμίσω ότι τα δικαιώματα των γυναικών βρίσκονται στη δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2017 και ε, είχαμε και οργανώσαμε ένα συγκεκριμένο σεμινάριο ε, ένα από τα βασικά επιτεύγματα είναι η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης και ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσχωρήσει στην ε, συνθήκη αυτή σύντομα. Ε, θα ήθελα τελειώνοντας να πω λίγα λόγια και μάλλον στο τέλος θα επανέλθω και θα μιλήσω για τα μέσα ενημέρωσης και για την ελευθερία του συνέρχεσαι. Γιατί τώρα πια δεν έχω χρόνο, νομίζω τελείωσε ο χρόνος μου. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, όταν συζητάμε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε καλέσει και το Συμβούλιο, την Ρουμανική Προεδρία. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι σημαντικά για τη Ρουμανική Προεδρία. Σας ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος, για το σχόλιο αυτό. Παρακαλώ να έχετε κατά νου το εξή. Αναφέρατε τη Ρουμανία ως ε, ε, μια ειδική περίπτωση Θα μεταφερθεί το σχόλιο στην Προεδρία και φαντάζομαι ότι μπορεί να θέλει να απαντήσει η Προεδρία. Και ας συνεχίσουμε με τη συζήτηση. Εκ μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Κουντρίτσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή ασχολείται με τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβίαση του κράτους δικαίου, διακριτική μεταχείριση, ρητορική του μίσους. Παραβίαση του διαχωρισμού της εξουσίας, έλεγχος του δικαστικού σώματος, προπαγάνδα στα μέσα ενημέρωσης, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ανησυχητικά. Και θα μπορούσε ε, η τάση αυτή να οδηγήσει και σε τρομοκρατία. Ο δήμαρχος του Γκτάνσκ έπεσε θύμα αυτής της τρομοκρατίας, θύμα του θεσμοποιημένου μίσους με το οποίο τα τελευταία τρία χρόνια στην Πολωνία είχαμε πάρα πολλές ε, εμπειρίες. Ανεκτικότητα, σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι ο Πάβελ Ανταμόβιτς δεν σκοτώθηκε ματέως. Αυτά πρέπει να έχουμε κατά νου όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα κράτη είναι κυρίαρχα και υπάρχει και η αρχή της επικουρικότητας, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να είναι πρόφαση για να μην τηρούμε τις βασικές αξίες. Μία τροπολογία μιλάει για την μικρή αποτελεσματικότητα του άρθρου 7 το Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει για την Πολωνία και την Ουγγαρία και για το αν παραβιάζουν τις διατάξεις της συνθήκης. Χάρη στον Φραντς Έγκελ, με τις καλές τροπολογίες, εκ μέρους του ΕΛΚ θέλω να πω ότι θα εγκρίνουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και σας παρακαλώ για άλλη μια φορά να τηρείτε το χρόνο σας, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Γκυγιόμ, εκ των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η αιτήσια έκθεση για την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να θεωρηθεί έκθεση ρουτίνα, αλλά αυτό δεν ισχύει. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το 2017 ήταν ένα βασικό έτος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτή η έκθεση σήμερα έχει κέρια σημασία. Χρειάστηκε κατά τις διαπραγματεύσεις να δείξουμε πολύ ισχυρή στάση για θέματα τα οποία είναι αδιαπραγμάτευτα. Το κράτος δικαίου Υπάρχουν πολλές απειλές κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, κατά των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ε, είναι μακρύς ο κατάλογος αυτών των παραβάσεων και πολύ συχνά οι χώρες άλλαζαν στάση. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθούν ε, τις τρέχουσες εξελίξεις με βάση το άρθρο 7 και να επιβάλλουν κυρώσεις αν αυτό είναι απαραίτητο. Όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών, η παρενόχληση των γυναικών απέκτησε σημασία και μεγάλο βαθμό χάρη στο κίνημα MeToo πρέπει τα κράτη-μέλη να εγγυώνται ίση πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό, σε δικαίωμα στην άμβλωση και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ισχύει σήμερα. Όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν για το σώμα τους με απόλυτη ασφάλεια. Η ομάδα μου προσπαθεί να τηρούνται αυτές οι βασικές αρχές Όσον αφορά την ε, μετανάστευση, τη μετανάστευση τα κράτη-μέλη ε, αρνούνται να οργανωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρά τις εκκλήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και καλούμε τα κράτη-μέλη για άλλη μια φορά να ε, δώσουν σημασία στη μεταρρύθμιση του κανονισμού του Δουβλίνου. Υπάρχουν θέματα όπως ο ρατσισμός, η ξενοφοβία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να εγγυηθούμε και τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και θα ήθελα να πω και χρόνια πολλά στην κόρη μου που είναι 18 ετών και ξέρω ότι με παρακολουθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ και χρόνια πολλά στην κόρη σας. Όταν έχει τόσο νέα μητέρα, θα είναι και μια θαυμάσια κόρη, ο κύριος Γιούρεκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, για το 2017. Στην Κίμζε, στη λίμνη Κίμζε, στη Βαβαρία, ένας, ε, μια νεαρή γυναίκα, ε, ε, πρόσφυγας, δολοφονήθηκε ως αποτέλεσμα μίσους κατά της χριστιανικής κοινότητας από κάποιον αιτούντα άσυλο. Η Σουηδία αρνήθηκε άσυλο την ίδια περίοδο αυτή σε μια νεαρή Ιρανή ηθοποιό που επίσης είχε γίνει χριστιανή κατά μέσο όρο, μία φορά κάθε 10 λεπτά υπάρχει κάποια ε, παραβίαση ε, κατά χριστιανικών ναών στη Γαλλία. Στη Γερμανία, ε, μία φορά κάθε τρεις μέρες. Δεν ήταν τόσο κακές οι επιδόσεις. Παράλληλα, κατά το 2017 οι ε, Θέμεν ε, βεβήλωσαν ε, ένα ναό. Η έκθεση αυτή μιλά για την ξενοφοβία, αλλά δεν μιλά για το μίσος κατά του χριστιανισμού. Είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να συζητηθεί. Και αυτή η σιωπή που επιβάλλεται για το μίσος κατά των χριστιανών αποδεικνύει έλλειψη σεβασμού. Κάτι το οποίο αυτή η έκθεση το επιτρέπει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, εκ μέρου των φιλελευθέρων, κύριος Μισελ. Κύριε Πρόεδρε, και το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και φέτος κάνει την έκθεση για το 2017 και κάνει έκκληση για να αναλάβουμε δράση κατά των παραδιάσεων των βασικών αξιών στα κράτη-μέλη. Αυτή η έκκληση είναι ακόμη πιο επίκαιρη σήμερα που πλησιάζουν οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουμε την επιλογή μεταξύ δύο ειδών Ευρώπης. Μια Ευρώπη δημοκρατική και φιλελεύθερη με τις οικουμενικές αξίες που αποτελούν τη βάση προστασίας των πολιτών όπως ίσχυσε από το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ή μια Ευρώπη που πηγαίνει αντίθετα στο ρεύμα της ιστορίας και που θεωρεί ότι η προστασία του κράτους δικαίου και η προστασία των μειονοτήτων είναι κάποια λεπτομέρεια που ε, ε, υποκύπτει στις αυταρχικές τάσεις ή σε κάποιες επιλεκτικές ηθικότητες. Οι πολιτικοί θα πρέπει να επιλέξουν το στρατόπεδο που θα ακολουθήσουν και αυτό να υπερασπιστούν έναντι των εκλογέων τους. Θέλω να τονίσω ότι είναι πλέον επίγον οι θύνοντες στα κράτη-μέλη να λάβουν ξεκάθαρα θέση υπέρ της δημιουργίας ενός μηχανισμού εποπτείας, όπως έχει ζητηθεί από την Sophie Intveld και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ένας μηχανισμός στον οποίο θα συμμετέχει και το Συμβούλιο και που θα επιβλέπει κάθε χρόνο την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη. Όταν δεν υπάρχει σαφής μαρτυρία των ελλείψεων στα κράτη-μέλη, θα μας λείπει ένα σημαντικό εργαλείο για να μπορέσουμε να υπερασπιζόμαστε τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κύριε Μισελ. Μισελ, μήπως... Βάλτε τα ακουστικά σας γιατί υπάρχει, λέει ο Πρόεδρος, ε, μία μπλε κάρτα την αποδέχεστε, προέρχεται από τον κύριο Γκόλνις. Yes. Oui. Ευχαριστώ και κύριε Μισελ και κύριε Πρόεδρε. Σύντομη η ερώτηση. Είστε πολιτικός Βέλγος εξέχων. Δεν εντυπωσιάζεστε που η χώρα σας, το Βέλγιο, έχει εδώ και κάποια χρόνια ως βασική αντιπολίτευση το Βλάμς Μπλοκ, το οποίο βρίσκεται την δικαστική απαγόρευση και εδώ στο κοινοβούλιο δεν ακούστηκε καμία φωνή διαμαρτυρία. Ο Μισελ. Όχι. Δεν με η υπογόρευση. γιατί παρανομή. Υιοθετεί συμπεριφορές αντισυνταγματικέ. Αυτή η παράδειξη κύριε Δόλνη. Τώρα λέγεται Flams Belang, όχι Flams Block. Ξέρω ότι είναι αδελφό σας κόμμα. Ε, τι να πούμε τότε. Πώς να κρίνουμε. Ούτε εσείς μπορείτε να κρίνετε τη στάση του Βελγίου έναντι ενός βεβαιωμένα φασιστικού κόμματος. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Μιράντα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πρώτα πρώτα. Μπράβο στον κύριο Τέρη για την εκθέση του. Αναδεικνύει αυτό που ονομάζουμε αξίες, αξίες και δικαιώματα. Αναλύεται η πραγματικότητα. Το 17 με τους ε, πρόσφυγες είδαμε τι γίνεται με τους ε, μετανάστες, με αυτούς τους πρόσφυγες, με αυτούς που έρχονται για να σώσουν την ζωή τους. Ήταν ε, ισοπεδωτική χρονιά, είχαμε τόσους νεκρούς στη Μεσόγειο. Να, ποια είναι η ιστορική μνήμη αλλά και για τα γυναικεία δικαιώματα, τα γενετήσια, τα αναπαραγωγικά, πολύ δύσκολη χρονιά. Ξέρω ότι βέβαια στην αποκή αυτό στη δεξιά πτέρυγα. Δύσκολη χρονιά για την ελευθερία έκφρασης, για τα ΜΜΕ, είχαμε συγκέντρωση των ΜΜΕ, είχαμε καταχρηστικές πρακτικές σε πολλά ΜΜΕ, Δυσμενεί διακρίσεις, ρητορική μίσους, να, τη διαπιστώσαμε ότι συνέβη αυτή τη χρονιά. Είδαμε τι απειλή φαίνεται από την κυρία Λεπέν και το Vox για την επόμενη θητεία. Η κυρία Βέρζια έχει το λόγο για την Γκουε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα πρώτα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους ε, σκιώδεις ηγητές. Ναι, σε αυτό το θεματολόγιο ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα δικαιώματα, τι γίνεται με το κράτος δικαίου ε, θα πρέπει ε, να είναι το θεμέλιο πάσης πολιτικής και όλα τα σχετικά, σχετικές παραβιάσεις θα πρέπει να τιμωρηθούν γιατί θέτουν εν το κράτος δικαίου και την δημοκρατία. Επίσης, είναι αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το μέτωπο με τα δημοσιομικά και τα οικονομικά. Να προσπαθήσει περισσότερο όμως ανεξαρτησία δικαιοσύνης, ελευθερία έκφρασης, ΜΜΕ, δικαιώματα των γυναικών, ε, ρητορική μίσους, με η γάγκρενα εξαπλώνεται. Ε, η, τα, τα, τα θύματα, τα ξυλαστήρια γίνονται οι μετανάστες. Είδαμε τη σουρελιστική προβληματική σε σχέση με τη συνάντηση κορυφής του Μαρακές και πόσες κυβερνήσεις υπονόμευσαν ε, αυτό το ομόφωνα εγκεκριμένο κείμενο του καλοκαιριού του 18. Έτσι η κατάσταση γίνεται πιο ευάλωτη. Η ιστορία θα είναι ανελέητη στην κρίση της σε σχέση με τους σήμερα κυβερνώντες. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Λαούρα Φεράρα για το EFDD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε χρόνο ε, βλέπουμε τι γίνεται ε, σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, βλέπουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι για την ισότητα ενώπιον του νόμου, της ελευθερίας, τα δικαιώματα, τι δυσμενεί διακρίσει, Όλα αυτά θα πρέπει να είναι το θεμέλιο κάθε δημοκρατικής δικαιοσύνη και κράτου δικαίου. Ε, άρα θα πρέπει να δούμε κάποια σημαντικά ζητήματα, ε, γιατί έχουμε διάφορα φαινόμενα τα οποία ξεπετάγονται σε κρατημέλη, ξενοφοβία, βία σε σχέση με τις γυναίκες, τους μετανάστες και τις μειονότητες. Ε, θα πρέπει να υπάρχει κράτος δικαίου και ελευθερία έκφρασης. Έχουμε επίσης και τη διαφθορά που και αυτή είναι μια απειλή για την ισότητα των πολιτών και να μην έχουμε διασπάθηση των ε, βρικοδοτήσεων των δημοσίων υπηρεσιών. Άρα χρειάζεται να στηθεί ένας μηχανισμός εποπτείας ευρωπαϊκός να βάλουμε φρένο στις καταπατήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι τώρα θα αντιμετωπίζουμε την ε, ε, ένδια, τη φτώχεια, ε, το πώς θα έχουμε εθνικά συστήματα ελάχιστου του εισοδήματος. θα πρέπει να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής ζωή, να δούμε πώς με την αγορά εργασίας θα μπορέσουμε να έχουμε ποιοτικό βιωτικό επίπεδο. Θα πρέπει επομένω από πλευρά οικονομική να θωρακίσουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να δούμε τι γίνεται με τις λιτότητες και τις ε, αγορές. Μα ε, να δούμε πώς ο κόσμος έχει κάποιες προσδοκίες που περιμένει από μας να τους βάλουμε στο επίκεντρο των πολιτικών μας. Χρειάζεται να υπάρξει κοινωνική ευημερία και να υπάρξει ε, όρων των δικαιωμάτων ε, ε, σεβασμός. Ευχαριστούμε. Ζήλστρα και το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε η πολιτική βία στην ε, Γερμανία και στην Πολωνία. Ε, νομίζω ο πρόεδρος ε, είπε ότι θα πρέπει να μιλάμε λιγότερο και να ακούμε περισσότερο ε, και πολλοί κάγχασαν. Εγώ το βρίσκω πολύ ανησυχητικό. Η βία κατά των πολιτικών δεν είναι μόνο σωματική, αλλά είναι και άλλη μορφή, διοικητική παραδείγματο χάρη. Αυτό πλήττει και το Κοινοβούλιο. Και όσον αφορά τις ε, εκλογές, ε, ελπίζω να αποκλειστούν πολίτες γιατί αποτελούν απειλή για την τάξη, την ελληνική τάξη πραγμάτων. Πρέπει λοιπόν να διερωτηθεί κανείς ε, κατά πόσον οι πολιτικές απόψεις ε, ε, δικαιολογούν τα πάντα, ακόμα και την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκόλμις είναι ο επόμενος ομιλητής. Γαλλικά. ναι, τα θεμελιώδη δικαιώματα απειλούνται στην Ευρώπη, αλλά όχι με τον τρόπο που περιγράφεται στην έκθεση. Η συσσόρευση νόμων περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης. Βλέπουμε ότι γίνεται κριτική του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και αυτά που είπε μόλις τώρα ο κύριος Μισελ. Μιλούσαμε για ένα ε, ειρηνικό κοινοβουλευτικό ε, κίνημα που εκπροσωπήθηκε στις εκλογές. Ο κύριος Μισελ όμως ε, με μια ρητορική μίσους μιλά για τους βουλευτές αυτούς ως αντισυνταγματικούς και θεωρεί δικαίωμα του δικαστηρίου να καταργήσει τα δικαιώματά τους. Υπάρχουν τα στερεότυπα της ομοφοβίας. Υπάρχουν εκατοντάδες πολιτικοί ε, ε, εχμάλωτοι στην Γερμανία. Η κυρία Ούρσουλα Χαβερμπέκ, 90 ετών, φυλακίστηκε στην ηλικία των 90 ετών ε, για θέματα ελευθερίας της έκφρασης. Οποία υποκρισία. Ο κύριος Σβόμποντα. Από την έκθεση αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το πρώτο μέρος που τονίζει το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται ε, ε, στο νόμο, αλλά η νομοθεσία δεν έχει ε, στην Ευρώπη τη δική της αστυνομία να την ε, υπερασπίζεται. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε το κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Δυστυχώς όμως η έκθεση αγνοεί εντελώς ε, τα θέματα μυσαλλοδοξίας έναντι των χριστιανών στην Ευρώπη. Και οι επιθέσεις κατά χριστιανών έχουν γίνει πάρα πολύ συχνές. Στην Αυστρία υπάρχει ένα νέο Ινστιτούτο που ερευνά το φαινόμενο αυτό. Το σύστημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων μας βασίζεται ε, στο σεβασμό του ατόμου και αυτό έχει χριστιανικές ρίζες. Χωρίς τις χριστιανικές ρίζες θα εκφυλιστεί το όλο σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από την κυρία Μαρία Γκραπίνη. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφοι, συμφωνώ μαζί σας Επαναλαμβάνω λοιπόν τώρα που βάλετε τα ακουστικά σας. Συμφωνώ ότι πρέπει να τηρούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μια και μιλήσατε για την Αυστρία. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για το ότι η Αυστρία ασκεί διακριτική μεταχείριση έναντι των παιδιών, μητέρων που δεν είναι ε, αυστριακές υπήκοοι, αλλά συνεισφέρουν στο ΑΕΠ τη Αυστρία, δουλεύοντα εκεί. já jsem eh, paní mluvil eh, o něčem úplně jiném já jsem mluvil o eh, diskriminaci. Εγώ μίλησα για κάτι εντελώς διαφορετικό. Μίλησα για τη διακριτική μεταχείριση κατά των χριστιανών στην Ευρώπη. Υπάρχει βέβαια, υπάρχουν πολλά είδη διακριτικής μεταχείρισης ε, που παραβιάζει το κράτος δικαίου και πολλοί μπορεί να επιβαρύνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα συμφωνούσα ούτε με αυτό το οποίο αναφέρεται. Ευχαριστώ. Θα ήθελα η κυρία Σοφή Ιντφελ να κάνει μια άλλη ερώτηση, παρακαλώ. έχετε όμως αυτή τη δεύτερη ερώτηση. Εντάξει, μα δεν κάνετε. Ναι, ευχαριστώ. Μιλήσατε για τους μαχητικούς αθειστές. Δεν καταλαβαίνω πώς δυσχεραίνουν τη ζωή των χριστιανών. Ίσως να είναι δυνατόν. Αλλά είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταρρεύσει αν δεν ε, συνεχίσει να βασίζεται στις χριστιανικές της αρχές. Αλλά αυτό που είναι κοινό δεν είναι περισσότερο ο διαφωτισμός και το κράτος δικαίου. Αυτή δεν είναι η βάση της κοινωνίας μας. Εντάξει, εγώ σέβομαι τις δικές σας ε, χριστιανικές ρίζες, αλλά αν δεν σέβεστε το γεγονός ότι άλλοι είναι άθεοι, πώς μπορούμε να συμβιώσουμε. Ε, Ευχαριστώ. Εγώ σέβομαι τις ε, πεπιθήσεις των πάντων, αλλά θέλω να τονίσω ότι ο σεβασμός μεταξύ των ατόμων είναι πολύ σημαντικός. Αν δεν υπάρχει όμως ε, σεβασμός με βάση τις χριστιανικές μας ρίζες, τότε αυτό θα οδηγήσει, και όπως ήδη συμβαίνει, σε μία ε, κατάρρευση. Ευχαριστώ για τις σαφεί απαντήσει σας. Τώρα ο κύριος Δίτμαρ Κώστα. Κώστα, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα βασικά δικαιώματα είναι διαρκή και κάθε πολίτης πρέπει να έχει τα προσωπικά του δικαιώματα τα οποία να μπορεί να τα απαιτήσει και ενώπιον, ενώπιον των δικαστηρίων. Αυτά είναι η βάση για την, ε, ε, το διαβασμό των εξουσιών, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Μόνο μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς είναι μια ανθρωπιστική κοινωνία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα δικαιώματα των μειονοτήτων πολύ συχνά δεν γίνονται σεβαστά για παράδειγμα, οι Ρώμα αντιμετωπίζονται με ρατσιστικές διακρίσεις και με εκνευρίζει ότι πάνω από 70 χρόνια μετά